Koleżanki i koledzy, συνάδελφοι, ξεκινά η συνεδρίασή μας και έχω κάποιες ανακοινώσεις να κάνω. Καταρχάς ανακοινώνω τη συνέχιση της διακοπής σας συνόδου που είχε διακοπή στις 17 Φεβρουαρίου.